Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι και συναδέλφοι Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι και φίλοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρόεδρο της Γεωργίας, τον κύριο Μιχαήλ Σακασβίλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Πρόεδρος επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχε έρθει και πριν από τέσσερα χρόνια εδώ στο Στρασβούργο, αλλά και στις Βρυξέλλες το 2004, αμέσως μετά την εκλογή του ως Πρόεδρο της Γεωργίας. Η σημερινή μέρα είναι ιδιάζουσα, γιατί σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια, Ελάμβανε χώρα η Επανάσταση των Ρόδων της ανέμακτης αυτής καμπής που άλλαξε την κατάσταση σε ολόκληρο τον Νότιο Κάφκασο και μάλιστα χάρη στην κατάσταση αυτή και χάρη στην αλλαγή αυτή ακολουθεί το δρόμο της ειρήνης, ένα δρόμο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διάλεξε πριν από 60 χρόνια. Θέλει αηφόρο ανάπτυξη, ευημερία και μια ελευθερία χωρίς και μάλιστα στο ο, κύριος Σακασβίλη έχει δεσμούς και με το Στρασβούργο. Ήταν και στο Κίεβο, σπούδασε και εκεί, αλλά και στο Στρασβούργο σπούδασε. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω στο Στρασβούργο γνώρισε την μέλουσα σύζυγό του. Οπότε για τον ε, κύριο Πρόεδρο το Στρασβούργο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Και μάλιστα η τελευταία, η τελευταία δεν ήταν καθόλου εύκολη για την Γεωργία. Γιατί απειλήθηκε η εδαφική ακυρεότητα της Γεωργίας και μάλιστα το Μάιο είχαμε εγκρίνει και σχετικό ψήφισμα καλώντας τη Ρωσία να τηρήσει τους ε, όρους της κατάπαυσης του πυρός και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το έδαφος της Γεωργίας. Πριν από τέσσερα χρόνια ο κύριος Πρόεδρος είχε πει σε αυτή την ίδια αίθουσα ότι οι Γεωργιανοί δεν είναι μόνο από τους αρχαιότερους λαούς της, Ευρωπαϊ... της Ευρώπης αλλά είναι ενθουσιώδεις υπέρμαχοι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πιστεύουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι η σωστή για τα διεθνή ζητήματα. Πιστεύω ότι και σήμερα ο ενθουσιασμός αυτός παραμένει αμύωτος. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στο δρόμο εκδημοκρατισμού της Γεωργίας, γιατί οι δημοκρατικές προδιαγραφές είναι πολύ υψηλές, της ελεύθερης αγοράς επίσης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά απαιτούν μεταρρυθμίσεις, συνταγματική αναθεώρηση, ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, του εκλογικού νόμου. Πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω όλα αυτά με τον πρόεδρο της Γεωργίας και συμφωνήσαμε ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά είναι απαραίτητη, γιατί έτσι θα διευκολυνθεί και η συνεργασία μεταξύ μας. Χαίρομαι γιατί η Γεωργία ξεπέρασε πολύ γρήγορα και την οικονομική κρίση. Βέβαια, σε αυτό συνέβαλε και η βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έτεινε χείρα βοηθεία. Και σήμερα η Γεωργία βρίσκεται και πάλι στο δρόμο τη ε, ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για μια σταθερή γεωργία και για μια ευημερούσα γεωργία. Αυτό μας ενδιαφέρει όμως για το σύνολο της περιοχής του Νοτιού Η γεωργία μπορεί να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, υπόδειγμα εφαρμογής του συστήματος της ελεύθερης αγοράς, του εκδημοκρατισμού, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εφαρμογής του κράτους δικαίου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας και μας ε, ενδιαφέρουν πολύ οι προτάσεις σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που βρίσκεστε ανάμεσά μας και σας δίνουμε το λόγο. Περιμένουμε με ζωηρό ενδιαφέρον την ομιλία σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σας καλωσορίζω. Ε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Η πρόσκλησή σας συνιστά τεράστια τιμή για τη χώρα μου και θα ήθελα ταπεινά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες τις πολιτικές ομάδες για αυτή την εξαιρετική ευκαιρία. Είχαμε την ευκαιρία να του συζητήσουμε πριν από τέσσερα χρόνια σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επανέρχομαι τέσσερα χρόνια μετά. Ελπίζω ότι η φορά αυτή να έχω καλύτερες επιδόσεις ε, στο άθλημα. Πάντως και πάλι παραμβάνω τεράστια τιμή. Έρχομαι εδώ να σα δώσω ένα μήνυμα ελπίδα και να αναλάβω μια επίσημη δέσμευση. Ήρθα εδώ να διατρανώσω ότι η ειρήνη δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη είναι δυνατή στην περιοχή μου και ότι χρειαζόμαστε την Ευρώπη για να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Επί αιώνες τα όρια του Καυκάσου ε, ήταν μυστήριο γεωπολιτικά, ένα παράδοξο. Μια περιφέρεια όπου ήταν ελεύθερα τα άτομα και οι ψυχές, αλλά οι πολίτες υποκαταστολή και καταπίεση. Οι πολιτισμοί ήταν ανεκτικοί, αλλά ε, οι κυβερνήσεις ε, δημιουργούσαν τεχνητές διαιρέσεις. Ο κόσμος ποτέ δεν, δεν έπαψε να αισθάνεται εκεί Ευρωπαίος, αλλά πάντα ε, κυριαρχούσαν ε, διάφορες ε, αυτοκρατορίες και έκανα την Ευρώπη μακρινό όραμα. Οι άνδρες και οι γυναίκες αγωνίζονταν για την ειρήνη, αλλά η ειρήνη αυτή φαινόταν κάτι το μακρινό. Θα πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Ε, θα πρέπει ε, να κυριαρχεί η ε, διαπραγμάτευση επί της ρητορίας του πολέμου. Κυρίες και κύριοι, σε όλες τις ταραγμένες γωνιές του κόσμου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σύμβολο ελπίδας. Η κατάφορη απόδειξη ότι καμία ειρήνη δεν αξίζει ένα πόλεμο ή πολιτικό κίνδυνο. Ακόμα και μέσω ερυπείων ε, ηγέτες Σαραλέη, ε, ε, κατάφεραν να τερματίσουν ε, τους πολέμους στην Ευρώπη και να προχωρήσουν σε ένα αξιοθαύμαστο πείραμα την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Το κοινοβούλιο σας δεν διαιρείται με εθνικότητες αλλά με πολιτικές ομάδες όπως τόσο εύγλωτα είπε το 1849 ο Βίκτορ Ουγκό στο Παρίσι στο Διεθνή Συνέδριο Ειρήνης. Και επιτρέψτε μου στα γαλλικά να παραθέσω αυτά που είπε ο Βίκτορ Ουγκό. Φέρθηκα κάποια μέρα που όλα τα έθνη της Υπήρου ε, χωρίς να χάσετε τις ε, ιδιαίτερες ε, αρετές σας και τα χαρακτηριστικά σας θα ενωθείτε σε μια Ευρωπαία αδερφοσύνη. Θα έρθει μια ημέρα που δεν θα γίνεται αντιπαράθεση στα πεδία των μαχών. Ε, θα έρθει μια μέρα όπου οι ε, βόμβες ε, θα αντικατασταθούν από τη καθολική ψηφοφορία από μια μεγάλη γερουσία κυρίαρχη που θα είναι για την Ευρώπη αυτό που είναι το κοινοβούλιο στην Αγγλία ιδιαίτερα στη Γερμανία και η Εθνοσυνέλευση στην Γαλλία. Οι περισσότεροι σύγχρονοι του Βίκτορος ο ο, θεωρούσαν ότι ήταν αφελής και ονειροπόλος και χρειάστηκαν πάνω από 100 χρόνια και δύο παγκόσμιοι πόλεμοι για να δικαιωθεί από την ιστορία. Κυρίες και κύριοι, έχει έρθει η ώρα να ακουστεί η ε, φωνή του Βίκτορ Σουγκό και στη δική μου περιφέρεια. Έχει έρθει ε, πλέον η ώρα αυτή η φωνή της αδελφοσύνης να ξεπεράσει τα σύνορα και τα μίση. Ε, είναι καιρός η ευρωπαϊκή ειρήνη να επεκταθεί και προς τον Κάφκασο. Και είναι δική μας ευθύνη ως πολιτικών ηγετών να ε, επινοήσουμε πρωτοβουλίες αραλές για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς πριν από 7 χρόνια έλαβε χώρα η Επανάσταση των Ρόδων και ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι προς την ευρωπαϊκή οικογένεια μιας ε, παλιάς ευρωπαϊκής χώρας, αγαπημένης μου ε, Γεωργία, 23 Νοεμβρίου 2003, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από κάθε προέλευση, ε, περιφέρεια, θρησκεία και κοινωνική ε, δύναμη έκανε Ειρηνική Επανάσταση. Δεν ε, υπήρξε καθόλου αντιπαράθεση, δεν έσπασε ούτε ένα τζάμι. Ήταν πραγματικά μια επανάσταση ε, που χαρακτήρισε ο οικόνομης του Λονδίνου ως επανάσταση της νοοτροπίας. Όπως γνωρίζετε, ε, ε, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης κατέρευσαν δύο Ευρώπες. Η Ευρώπη του κράτους δικαίου και η Ευρώπη του φόβου. Ο διχασμός που επικρατούσε ξεπεράστηκε επικράτησε η Ευρώπη του Βάκλαρ Χαβέλ απέναντι στην Ευρώπη του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Πριν από 7 χρόνια Κυρίες και κύριοι, η Γεωργία ήταν επίσημα ε, ανεξάρτητη χώρα, αλλά ε, παρόλα αυτά ε, επικρατούσε ο φόβος και το μίσος. Η σοβιετική νοοτροπία δεν είχε καταπέσει, η Σοβιετική Ένωση παρέμενε ε, στο νου και ε, στην καρδιά ε, των πολιτών. Μόνο μια επανάσταση νοοτροπίας θα μπορούσε να αλλάξει τις κοινωνίες μας. Αυτό το μήνυμα φέραμε εμείς οι Γεωργιανοί στην περιοχή και αυτό γέννησε τόσο μεγάλο θυμό μεταξύ των νοσταλγών της αυτοκρατορίας. Αυτό όμως το μήνυμα έκανε τη Γεωργία ένα εργαστήριο ιδεών όλοι οι ενεχόμενοι στην επανάσταση των Ρόδων, ε, κόμματα της αντιπολίτευσης, φοιτητέ, κοινωνία των πολιτών είχαν ένα όραμα να αναστήσουν τη χώρα που είχε καταβληθεί από τη διαφθορά και τη Σοβιετική εποχή και να την κάνουν πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, η Σοβιετική Ένωση βασιζόταν σε μια αρχή, διέρη και βασίλευε με τεχνητές ε, διαιρέσεις και αντιπαλότητες σε κάθε τομέα της κοινωνίας πολιτικής, σε διάφορες ομάδες θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνοτικές ε, ήταν πραγματικά το κράτος του φόβου, του μίσους και της χειραγώγησης. Αυτό εξηγεί γιατί οι πρώην κομμουνιστές ηγέτες τόσο εύκολα γίνονται εθνικιστές και στα Βαλκάνια και στον Κάφκασο και στην Ανατολική Ευρώπη και στη Ρωσία. Πριν από 7 χρόνια η Γεωργία ήταν ακόμα διαιρεμένη σε απομονωμένες κοινότητες ε, που η μία φοβόταν την άλλη και απέριπτε τις μειονότητες στο κράτος. Γι' αυτό το πρώτο μας καθήκον ήταν να αγκαλιάσουμε την ε, πολυπολιτισμική διάσταση και τις διαφορές. Παντού ε, και μέχρι τα πανεπιστήμια και ε, τις δυνάμεις ε, της τάξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σοβιετική Ένωση είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό τον πλήρη συγκεντρωτισμό. Γι' αυτό εμείς ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα αποκέντρωσης και στις υποδομές και ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ως αποτέλεσμα, περιφέρειες που στο παρελθόν ήταν ε, εγκαταλελειμμένες ε, έγιναν πραγματικά ανθούσες περιοχές ανάπτυξης. Μέχρι την επανάσταση των Ρόδων, όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν από τον Πρόεδρο με μια κάθετη, όπως γνωρίζετε, δομή, χωρίς αυτονομία στις περιφέρειες και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντίθετα, ε, ε, πέρσι το Μάιο ε, εξελέγει για πρώτη φορά άμεσα ο δήμαρχος της Τυφλίδας και ελήφθη απόφαση να μετακατασταθεί το συνταγματικό δικαστήριο στο Βατούμι και το κοινοβούλιο στο Κουτάισι. Η πρώτη μας απόφαση, λοιπόν, το πρώτο βήμα ήταν να διαλύσουμε την ΚΑΓΕΜΠΕ να απολύσουμε το σύνολο των αστυνομικών και των ε, φοριακών και των τελωνιακών και να ανοίξουμε την οικονομία μας και την παιδεία μας ένα ήταν το σύμβολο ε, στο όραμα αυτό. Ε, εκτός από τη σημαία της Γεωργίας, σε κάθε επίσημο κτίριο εγκαταστήσαμε την Ευρωπαϊκή Σημαία για να δείξουμε ε, προς τα πού θέλουμε να φέρουμε τη Γεωργία με τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως έκανε και σφάλματα και είχε και ελλείψεις η επανάστασή μας. Βεβαίως κάναμε και εμείς λάθη. Αλλά ε, ως ο, μέγας εφευρέτης του κοσμολιτισμού στην Ευρώπη και ένας από τους αγαπημένους μου φιλοσόφους, ο Ιμάνολ Κάντ έγραψε για τη Γαλλική Επανάσταση, δεν μπορεί να είσαι έτοιμο, να γίνει ελεύθερο, μέχρι να είσαι πραγματικά ελεύθερο. Τι εννοούσε ο Καντ κύριε και κύριοι, ότι δεν μπορείς ένα εγχειρίδιο να διδαχθεί εκ των προτέρων πώ να κυβερνά ή πώ να φέρεσαι σε συνθήκε ελευθερίας. Αυτά τα μαθαίνει μόνο από τι ίδιε τι επιτυχίε και τι αποτυχίε. σου. Είχαμε και αποτυχίε και διδαχθήκαμε από αυτέ, αλλά είχαμε και εκπληκτικέ επιτυχίε. Η Παγκόσμια Τράπεζα ξεχώρισε τη Γεωργία ως υπαριθμό ένα οικονομικό μεταρρυθμιστή παγκοσμίω τα τελευταία πέντε έτη. Και τώρα βρισκόμαστε στη 12η θέση στον κόσμο ε, ε, ως ε, χώρα για ευκολία επιχειρήσεων και υπαριθμό ένα στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην Σοβιετική Ένωση κάποτε ήταν το επίκεντρο της μετασοβιετικής μαφίας η Γεωργία, αλλά έχει κάνει τεράστια πρόοδο από το 2004 στο 2009, σύμφωνα με τη διεθνή διαφάνεια. Στην κατάταξή της η Γεωργία ανέβηκε 70 θέσεις. Και αντίθετα έπεσε και η Ρωσία κατά 70 θέσεις και συναντηθήκαμε κάπου στη μέση ε, ε, ανεβαίνοντας, τους χαιρετήσαμε ενώ κατέβαιναν αυτοί. Ε, αξιολογώ αυτή την κατάταξη γιατί δείχνουν πραγματικά πόσο βαθιά ήταν η μεταρρύθμιση στη χώρα μου και η επανάσταση της νοοτροπίας που σας ανέφερα προηγουμένως. Οι γεωργιανοί πολίτες σταμάτησαν να θεωρούν τη χώρα τους ως μια μετασοβιετική χώρα, το κράτος ε, δηλαδή. Το βλέπουν, το κρίνουν και συχνά το ε, επικρίνουν ως Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Αυτές οι αλλαγές ξεπερνούν βεβαίως τα κόμματα και ε, τους ηγέτες της Επανάστασης των Ρόδων. Κανείς ε, δεν ε, έχει διοκτησία αυτό το γεγονός και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει, ούτε εμείς ούτε κανένας άλλος. Και ακολούθησε κάτι το εκπληκτικό, ότι συστηματικά οι θεσμοί είναι πιο δημοφιλείς από ότι τα κόμματα οι ηγέτες. 86% σήμερα ε, χέρι εμπιστοσύνη ε, η αστυνομία, ενώ στο παρελθόν ήταν 5%. Το ίδιο για του άλλου θεσμού ισχύει. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ εύγλωτο και δείχνει ότι ε, όταν οι θεσμοί είναι πιο δημοφιλεί από του ηγέτε, η χώρα πάει καλά, πάει στη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίω έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε και είμαστε περισσότερο από ποτέ προσιλωμένοι στι μεταρρυθμίσει. Γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία είναι πάντα ε, ένα έργο ε, εξελισσόμενο. Κυρίες και κύριοι, δεν χάρηκαν όλοι από αυτή την αλλακτική δημοκρατική πορεία. Γνώρισε στεναρία ε, αντιπολίτευση και αντίσταση μεταξύ κύκλων αναθεωρητικών που νοσταλγούσαν ε, το παρελθόν και θεώρησαν τη μεγαλύτερη καταστροφή του 20ου αιώνα την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ε, ε, επέβαλαν εμπάργο πλήρες στη χώρα μας το 2006, έδιωξαν τους πολίτες μας και τελικά εισέβαλαν το 2008. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, οι δυνάμεις αυτές κατέχουν το 20% της επικράτειάς μας σε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Συμφωνίας Κατάπαυσης του ε, πυρός της 12ης Αυγούστου ε, που επετεύθη χάρη στις προσπάθειες του καλού μου φίλου ε, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζή που τότε προέδρευε. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ είναι 500.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι και οι πρόσφυγες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις αιστείες τους γιατί κάποιοι που έχουν παλιωμοδίτικες ιδέες αυτοκρατορικές θεωρούν ότι τον 21ο αιώνα μπορούν να κάνουν εκστρατείες εθνοτική κάθεσης και μπορούν να στείλουν νέα τύχη του Βερολίνου στη χώρα μου. Πώς απαντήσαμε εμείς αυτή την εισβολή. Ε, ε, Πλήρω εφαρμόσαμε τη Συμφωνία Κατάπαυση του Πυρός και πέρα από τις υποχρεώσεις μας, ε, παρόλο που ε, η Ρωσία ε, ανήθηκε. Πέρυσι τον Αύγουστο, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης, ο Hans Χάμπερ, γερμανός πολίτης, επένεσε τη στάση της Γεωργίας, τη συγκράτησή της, ως επικοδομητική μονομέρεια. Έχουμε άρματα μάχης και πυράβλους που σταθμεύουν 50 χιλιόμετρα από την Τυφλίδα ότι ε, θέλουν να μας δείξουν ότι είναι πολυτέλεια η δημοκρατία και η ελευθερία ε, και ορισμένοι ζητούν να κλείσει αντιπολίτευση και να ενωθεί η κοινωνία, να προχωρήσουμε στην ενότητα της κοινωνίας. Κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Κυρίε και κύριοι, δημιουργούμε μια δημοκρατία με το πιστόλι στο πρό... στον πρόταφο. Μπροστά από το σιδηρούν παραπότασμα που έκτισαν οι δυνάμει κατοχή γύρω από την περιοχή τη Απχαζία, στη μικρή παραθαλούση απόλυτη Ανάκλεια, που ήταν ε, μια ε, no man's land πριν από κάποια χώρα, δημιουργείται ένα τουριστικό θέρετρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με πανέμορφα ξενοδοχεία και αμμουδερέ παλααλίε. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε και να περιμένουμε να επιληθεί η κατάσταση και μόνο τότε να αρχίσουμε με να οικοδομούμε όταν δεν θα τρέμει πλέον το έδαφο, θα είναι πιο σταθερό και λιγότερο επικίνδυνο. Η φιλοσοφία μα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Κατασκευάζουμε κτίρια όχι γιατί βρίσκονται σε στερεό έδαφο, αλλά γιατί κατασκευάζοντα τα θα κάνουμε πιο στερεό το έδαφο. Στην Ανάκλεια ξεκίνησε μια νέα φάση ανάπτυξη το 2005, αφότου καταστράφηκε ολοσχερός ε, η πόλη ε, δύο φορές, το 1993 και το 1998. Το 2008 και πάλι καταστράφηκε ολοσχερός ε, από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων. Καταστράφηκαν και δισκοτέκ, καφετέριες, ξενοδοχεία και Λίγες εβδομάδες αργότερα ξεκίνησαν εκ νέου κατασκευέ. Ένας μεγάλος ποιητή, ένας από τους μεγάλους διάσημους Ρώσους αντιφρονούντες, ο Αλεξάνδρ Γκάλιξ, ένας από τους οκτώ ήρωες που διαδήλωσαν στην Κόκκινη Πλατεία το 1968 κατά της εισβολής στην Πράγα, έγραψε αυτή τη μεγάλη φράση. Λαμπρή και υπεράφωνη χώρα απαντά στη λάσπη με ένα χαμόγελο. Έγραψε για τη Γεωργία Μία ακόμα υπέροχη φράση, θα την πω και πάλι στα ρωσικά. Που χονδρικά σημαίνει ότι η υπέροχη χώρα μας απαντά στη λάσπη με χαμόγελο. Last time. Την τελευταία φορά που επισκέφθηκα την Ανάκλεια, είδα μια σειρά από δισκοτέκ πάρα πολύ ζωντανέ, όπω θα βλέπετε σε οποιαδήποτε άλλο μέρο τη Ευρώπη, όπου νέοι άνθρωποι χόρευαν όπω θα το έκαναν στην Ήμπιθα ή στο Σαντροπέ. Η μόνη διαφορά ήταν ότι στην τελευταία δίσκο που πήγαμε, στην 18η, ήταν η τελευταία και 100 μέτρα από εκεί υπάρχει ένα τείχο που έχουν ανυψώσει οι δυνάμεις κατοχής και εκεί βρίσκεται ο στρατός κατοχής. Να σας ρωτήσω το εξής. Και μετά και 100 χιλιόμετρα είναι σκοτεινά τα, τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει τίποτα πιο παράλογο από ένα νέο τείχος του Βερολίνου σε μια ε, παραλία. Κυρίε και κύριοι, με λίγα λόγια καταλαβαίνουμε ότι η ειρήνη είναι το υπέρτατο συμφέρον μα και ε, είμαστε πεπισμένοι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την ειρήνη. Αν διακυβεύσουμε την ειρήνη, ουσιαστικά διακυβεύουμε όλα όσα επιτύχαμε και όλα όσα θέλουμε να επιτύχουμε στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα εδώ να σας ανακοινώσω ένα νέο βήμα στην πολιτική μας της επικοδομητικής μονομέρειας. Είμαι εδώ για να αναλάβω μια πρωτοβουλία που ελπίζω ότι με τη βοήθειά σας θα ε, αμβλύνει τις εντάσεις και θα επιτρέψει να ξεκινήσουν οι σοβαρές διαπραγματεύσεις. Πριν έρθω το σκέφτηκα πολύ σοβαρά, διαβουλεύτηκα και τους φίλους μας, τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ε, συμμάχους, ανθρώπους στην περιοχή και η γεωργιανή κυβέρνηση ήδη θεωρεί ότι δεσμεύεται από την ε, Συμφωνία Κατάπαυσης Πυρός της 12 Αυγούστου και θεωρεί πάντα ότι αυτή η κατάπαυση πυρός απαγορεύει τη χρήση βίας. Αλλά για να αποδείξουμε ότι η Γεωργία δεσμεύεται πλήρως ε, σε μια ειρηνική επίλυση στη διαμάχη της με τη Ρωσική Ομοσπονδία, Λαμβάνουμε σήμερα τη μονομερή πρωτοβουλία να δηλώσουμε ότι η Γεωργία δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ βία για να αποκαταστήσει την εδαφική της ακαιρεότητα και κυριαρχία και για να αποκαταστήσει τον έλεγχό της στις κατεχόμενες περιοχές. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ειρηνικά μέσα για να μπορέσουμε να έχουμε επανένωση της ε, περιοχής ακόμα και αν η Ρωσική Ομοσπονδία αρνηθεί να αποσύρει τα στρατεύματά τη, ακόμα και αν οι στρατιωτικές οργανώσεις που πρόσκυνται σε αυτήν ε, συνεχίσουν να κάνουν κατάφορες παραβιάσεις η Γεωργία θα ε, διατηρήσει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και θα σταματήσει τις διαπραγματεύσεις. Θα αποστείλω σχετικέ επιστολέ στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Γενικό Γραμματέα τη ΟΑΣΕ και φυσικά στην ε, ε ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντα σαφώ ότι δεσμευόμαστε να μην χρησιμοποιήσουμε δύναμη για να αποκαταστήσουμε τον έλεγχο στην παρανέμω ε, διαιρεμένη χώρα μα, ούτε κατά των κατοχικών δυνάμεων, ούτε κατά των τοποτηρητών, ακόμα και αν η χάρτα των Ηνωμένων Εθνών μα το επιτρέπει. Η δέσμευσή μου εδώ ενώπιον σα αποτελεί μονομερή δήλωση μια χώρας βάσει του διεθνού δικαίου. Αυτή η πρωτοβουλία κυρίες και κύριοι Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη για μια χώρα η οποία είναι κατεχόμενη μερικώ και έχει 500.000 εσωτερικώ εκτοπισμένου και πρόσφυγε. Συνεχίζει και επεκτείνει την πολιτική μα τη επικοδομητική μονομέρεια. Κυρίε και κύριοι, είμαι διατεθειμένο να κάνω ένα ει βάθο και εξαντλητικό διάλογο με τον ε, Ρώσο εταίρο μα. Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στι συζητήσει τη ε, Γενέβη, ελπίζοντα ότι η σημερινή μα δέσμευση θα πείσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει ε, να μπλοκάρει χάρη τις διαπραγματεύσεις, αλλά χρειαζόμαστε ε, την έναρξη και του πολιτικού διαλόγου. Και για να συμβεί κάτι τέτοιο, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να διασαφηνίσει στους Ρώσους ηγέτες ότι η κατάσταση ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για να τους πιέσουμε να συζητήσουν μια συμβιβαστική λύση, είναι σημαντικό να δηλώσουμε πώς έχει η κατάσταση επιτόπου. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε το ρωσικό ε, ε, στρατιωτικό κτίσμα εντός των διεθνών συνόρων της ε, Γεωργίας να θεωρείται παράνομη κατοχή ε, κυρίαρχης χώρας. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένε Πολιτείες το έχουν δηλώσει δεν είναι στρατιωτική κατοχή, τι είναι στρατιωτικό τουρισμό όπου έχουν έρθει άρματα και στρατεύματα και έχουν ε, κατασταθεί σε ε, συγκεκριμένο ογκάθι. Έχουν απελαθεί εκατοντάδες χιλιάδες γεωργιανοί πολίτες από τα κατεχόμενα εδάφη και αυτοί θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως εθνοτική κάθαρση. Εάν δεν καταγγείλουμε αυτή την εθνοτική κάθαρση, γιατί να σκεφτούν καν οι δυνάμεις κατοχή να τους επιτρέψουν να επιστρέψουν στις αιστείες τους και στα χωριά τους και τις πόλεις τους. Κυρίες και κύριοι, αν το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια, η αλήθεια είναι πάντα το πιο στέρεο θεμέλιο της ειρήνης. Η επικοδομητική μας μονομέρεια και η δέσμευση που μόλις έκανα ενώπιον σας δεν θα έχει τις αναμενόμενες επιπτώσεις αν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας δεν πούν την αλήθεια. Εάν δεν μπείτε εσεί την αλήθεια, Ποιο θα την πει. Ήρθα εδώ σήμερα για να σας πω ταπεινά ότι εμείς και όλη η περιοχή εξαρτώμεθα από εσά. Κυρίες και κύριοι, η περιοχή μας έχει γνωρίσει πάρα πολλούς πολέμους στην πρόσφατη ιστορία. Ήγηκε η ώρα να παραφράσω για άλλη μια φορά τον Βίκτορ Ουγκό και να ε, αντικαταστήσουμε τα κανόνια με στρογγυλές τράπεζες. Η περιοχή μα έχει τη δική τη Βαρσοβία, το δικό τη Κόβεντρι, το δικό τη Οραντούρ Σουργκλάν και πρέπει από κοινού να προχωρήσουμε την, ε, μέσω της απόρριψης του πολέμου και της καταστροφές. Δεν θα πρέπει να έχουμε μια άλλη ε, γκρόσνη, μια πρωτεύουσα 400.000 κατοίκων που εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ήγηκε η ώρα να πούμε ότι δεν θα πρέπει να ε, εκδιώκονται άνθρωποι από τις αιστείες τους, ούτε να απολέσονται βάσει της εθνικότητάς τους, ε, ε, των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων ή της καταγωγής τους, όπως συνέβη με τη χώρα μου και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ με τη ρωσική ηγεσία, ε, ώστε οι συνέπειε του πολέμου να αναστραφούν και να καθοριστούν οι προποθέσει για την ειρήνη. Τύχη όπως αυτά που διαιρούν τη Γεωργία δεν θα πέσουν μέσω όπλων ή από αλλά από τη δέσμευση των πολιτών να δημιουργήσουν μια ελεύθερη ενωμένη χώρα και από τη δέσμευση τη παγκόσμια κοινότητα να ενισχύσει το διεθνές δίκαιο. Και αυτή τη φιλοδοξία δεν θα την ε, απαρνηθούμε ποτέ. Δεν θα απαρνηθούμε ποτέ το δικαίωμα να έχουμε μια ειρηνική διαβίωση με τα ένομα μέσα. Καμία πρώην Σοβιετική Δημοκρατία δεν έχει αναγνωρίσει τη διάλυση της Γεωργίας. Μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι παλιοί καιροί έχουν παρέλθει προπολού. Δείχνει ότι τα πρώην ε, κατεχόμενα έθνη των Σοβιετικών καιρών έχουν γίνει πλέον ισχυρά ανεξάρτητα κράτη που καθορίζουν τα ίδια τις πολιτικές τους. Κανένας ε, δεν θα επιστρέψει στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Κυρίες και κύριοι, η περιοχή μας έχει κάνει την επιλογή της και ξεκίνησε ένας πόλεμος για να σταματήσει αυτή την κίνηση, αλλά τα τάγκς δεν μπορούν να αντιστρέψουν την αίσθηση της ιστορίας και είναι καιρό να σταματήσει αυτή η επώδυνη δαμόκλειες πάθη του υπεριαλισμού ε, με ειρηνικό τρόπο. Σας καλώ λοιπόν, ε, καλώ και τους Ρώσους ηγέτες να κάνουν την επιλογή αυτό για το μέλλον. Θα μπορούσαν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ε, συνεχώς για την αέναη αλλαγή της περιοχής μας, δεχόμενη τις χώρες ως εταίρους και όχι ως επιτελείς. Θέλουμε να έχουμε μια Ρωσία ως εταίρο και όχι ως εχθρό. Θα πρέπει να σέβεται η Ρωσία το διεθνές δίκαιο και αυτό φυσικά ε, ε, συχνά βασίζεται και στην ε, τήρηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ υποστήριξη από όλους τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ηγέτες για να συμμετέχει η Ρωσία σε μια επικοδομητική σχέση. Η σύραξή μας δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να αλλάξει την οτροπία μεταξύ των λαών μας. Θέλω να πω στους ρώσου ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στη Γεωργία ως εταίροι, ως τουρίστες, ως φοιτητές, ως επιχειρηματίες, ως δημοσιογράφοι ή απλώς ως φίλοι, αλλά όχι ως κατοχικέ δυνάμεις. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σταματήσω να ολοκληρώσω αυτή την ομιλία με μια δήλωση του Προέδρου της πρώτης Γεωργιανής Δημοκρατίας, της Νοέ Τζορντάνια. Όπως θα γνωρίζετε, η Γεωργία ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατική Δημοκρατία το 1918. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα για το Σύνταγμά μα προέκυψαν από εκεί. Λίγε μέρε αργότερα, πριν ε, εισβάλλει ο Ερυθρός στρατό στη Γεωργία, ο Ζορντάνη εξήγησε ποια είναι η ευρωπαϊκή μα ε, επιλογή. Αυτό που παίρνουμε από το πολιτιστικό φάσμα των ευρωπαϊκών εθνών, 2.000 εθνικού πολιτισμού, δημοκρατικού συστήματο ε, και φυσικού πλούτου. Εμείς ζητάμε από τη Ρωσία να συμμετέχει και θέλουμε η Ρωσία να συμμετέχει μαζί μα και να προχωρήσουμε προ την Ευρώπη. Σήμερα είναι εδώ ένας άλλος Γεωργιανός Πρόεδρος, αποστέλει το ίδιο μήνυμα αγάπη για τα ευρωπαϊκά ιδανικά και Αξία. Σπάνια δίνεται σε ένα έθνο ε, στην ιστορία το, η ίδια δυνατότητα δύο φορέ. Ήρθα εδώ σήμερα για να σα πω ότι θα δράξουμε την ευκορία και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα προκειμένου να επιτύχουμε το ευρωπαϊκό μα μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή η ομιλία και η παρουσίαση ήταν πολύ σημαντική για όλους μας, αλλά ήταν εξίσου σημαντική για την μελλοντική διάσκεψη κορυφής της ΟΑΣΕ που θα γίνει στην Άστονα στο Καζακστάν σε μία εβδομάδα, την 1η και Δευτέρα Δεκεμβρίου. Και φυσικά ήταν κέρια σημασίας ε, η, ε, η δυνατότητα αυτή για την περιοχή σας και για την συνένωση του, της περιοχής του Βορείου Καυκάσου και του Νοτιού Καυκάσου γιατί γνωρίζουμε ότι η περιοχή αυτή έχει θρέψει πολύ γενναίους άνδρες αλλά ταυτόχρονα και συνετούς και το κουράγιο, η τόλμη και η σύνεση θα πρέπει να βαδίζουν παράλληλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.